Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, τις, ε, είχαμε κάποια καθυστέρηση ε, για να έρθουν όσοι αντικαταστήσουν ε, τα μέλη για την ψηφοφορία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη αν δεν υπάρχει ένσταση ή κάποιος έχει ένσταση για τη σημερινή ημερήσια διάταξη. Έχει να πει κάτι. Δεν βλέπω να θέλει κανείς το λόγο. Οπότε μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Πάμε στην σημείο 2, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων. Σχεδίο πρακτικών του συνε... της συνεδρίασης 4ης 5ης Σεπτεμβρίου θα βρείτε στα έγγραφά σας. Υπάρχουν παρατηρήσεις για το πρωτόκολλο αυτό, για τα πρακτικά αυτά. Δεν βλέπω. Προτείνω λοιπόν να εγκρίνουμε τα πρακτικά αφού δεν, υπάρχουν, δεν υπάρξει ένσταση κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, στο τέλος της συνεδρίας θα θεωρηθεί ότι τα πρακτικά έχουν εγκριθεί. Πάμε στι ανακοινώσει τη Προέδρου, τρίτο σημείο. Πρώτα απ' όλα για τη διερμηνία. Σήμερα έχουμε διερμηνία για τι ακολουθέ γλώσσε: γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, τσέχικα, ουγγρικά, λιθουανικά, λετωνικά, πολωνικά, σλοβακικά, σλοβενικά, βουλγάρικα, ρουμάνικα και κροατικά. να ευχαριστήσω θερμό του διερμηνεί σήμερα για την εργασία του. Για το web streaming τώρα να σα θυμίσω ότι η συνεδρίαση αυτή μεταδίδεται με web stream. Μπορεί να τη δει οποιοδήποτε από οπουδήποτε. Αποφάσει τη 24η Σεπτεμβρίου των συντονιστών. Οι αποφάσει των συντονιστών τη 24η Σεπτεμβρίου του 2019 που εστάλησαν σε όλα τα μέλη της κάλτης της 25 Σεπτεμβρίου μέσω email θα πρέπει να ελεγχθούν και στις, ε, μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου έπρεπε να υποβληθούν όλες οι συνστάσεις. Θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί. Οπότε πάμε στην ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε εδώ πρώτα απ' όλα το σχέδιο γνωμοδότησης για το Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Η Πέτρα Κάμερεβερτ ήταν η συγγήτρια. Να ρωτήσω την Πέτρα Κάμερεβερτ αν θέλει να πάρει το λόγο. Ε, να είστε σύντομοι παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θέρμα όλους τους και ηγέτες και τη γραμματεία κυρίως και τους ε, συνεργάτες μας ε, για την εξαιρετική συνεργασία και την επικοδομητική του συμβολή, στη πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Βρίσκονται όλοι εδώ. Έχετε τις κάρτες σας για την ψηφοφορία. Δεν βλέπω να λέει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ας κάνουμε έναν έλεγχο και μετά να περάσουμε απευθεία στην ψηφοφορία. Πάμε συμβιβαστική 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά αποχές να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Electronic check, please. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 17 προς 12. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές δεν βλέπω καθαρά πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν άπαντες πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία 8 αποσύρθηκε τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογ... Ε, συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε σε βιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία επί του συνόλου του κειμένου ηλεκτρονική άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 25 υπέρ, 4 κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια στην Πέτρα Κάμερεβερτ για την έκθεση. Dann kommen wir zu Tagesordnung. Πάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης να προσπαθήσουμε για μια φορά να εκλέξουμε τον τέταρτο ή την τέταρτη αντιπρόεδρο για την Επιτροπή μας ε, με ενημέρωσαν ότι τα ακόλουθα μέλη θέλουν να λάβουν ε, μέρος στην ψηφοφορία ως αναπληρωματική κυρία Μπεντζουμέρ αντί για τον κύριο Ζαγοράκη και η Ντεβίντλερ για τον κύριο Φρανκόφσκι και, κυρία, και ο κύριος Έμπαν Καρθία Ντελάνκο αντικαθίσταται, αντικαθίσταται ο Παρακαλώ, κυρία Ζεμπού. Συγγνώμη, ευχαριστώ. Θέλουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ένα λεπτό να βάλω τα ακουστικά, λέει πρόεδρο. Επαναλαμβάνω, θα θέλαμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για αυτό το σημείο, παρακαλώ. Ε, μυστική, συγγνώμη, μυστική. Πολύ ωραία. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ε, ότι θα έχουμε μια αλλαγή για τους... Αν υπάρξουν άλλες αλλαγές, ε, να υπάρξει ενημέρωση για τους αναπληρωτές, για τους αναπληρωματικούς. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει απαρτία. Είναι, είμαστε περισσότεροι σήμερα σαφώς, οπότε ε, υπάρχει, διαπιστώνεται απαρτία. οκτώ είναι το ελάχιστο. Ποιο, ποιοι είναι είναι υποψήφη για Αντιπρόεδρη η κυρία Ζορκοβά. Παρακαλώ. Θα ήθελα να προτείνω τον συνάδελφο Ανδρέα Μποτσικό ως Την Αντρέα Μποτσικό ως αντιπρόεδρο. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες προτάσεις. Δεν βλέπω να προτείνει κάποιος κάποιον. Αφού έχουμε μια υποψήφια λοιπόν προτάθηκε από τους πράσινους να έχουμε μυστική ψηφοφορία, οπότε να σας ρωτήσω υπάρχουν άλλοι οι οποίοι το ζητούν αυτό, γιατί χρειαζόμαστε τουλάχιστον 7 μέλη για να γίνει ε, μυστική ψηφοφορία. Και οι αριστεροί λένε ναι, οπότε το έχουμε πάνω από 7 μέλη λοιπόν. Είπαμε τώρα ότι ε, διαπιστώνουμε ότι η κυρία Μπότσκο είναι πλήρες τακτικό μέλος. Ε, οι δηλώσει της για τα οικονομικά της συμφέροντα και η, και η δήλωσή της για την ε, συμμόρφωση με τον κώδικα διοντολογίας έχουν δοθεί. Θέλω να ζητήσω στην, την κυρία υποψήφιο αν συμφωνεί με την πρόταση αυτή. Όπως είπαμε θα κάνουμε μυστική ψηφοφορία, οπότε τώρα μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Από τους παρόντες, ε, από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, μήπως δεν έχει την κάρτα ψηφοφορίας. Έχετε όλη τις κάρτες ψηφοφορίας. Να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία για να δούμε ότι λειτουργούν οι συσκευές. Ας ψηφίσουμε λοιπόν ε, τον Πλάσιο Ντομίνγκο αν θέλουμε να γίνει μέρος της Επιτροπής μας. Με το πράσινο κουμπί ψηφίστε υπέρ και με το κόκκινο κατά. Και όποιος θέλει να αποσχεί μπορεί να πατήσει το μεσαίο λευκό κουμπί. Ας ψηφίσουμε λοιπόν τον Πλάσιο Ντομίγο. Ich Ψήφισαν άπαντες. Ωραία, κλείνουμε την ψηφοφορία. Ο Πλάσιο Ντομίγκα λοιπόν με 18 ψήφους εξελέγει Μετά από αυτή τη δοκιμαστική ψηφοφορία διαπιστώνουμε λοιπόν ότι λειτουργούν όλα τα μηχανήματα οπότε μπορούμε να περάσουμε στην πραγματική ψηφοφορία. Χρειάζεται πάντα να ελέγχουμε για να μην ε, είναι άκυρη η ψηφοφορία. Με το πράσινο λοιπόν κουμπί ψηφίζουμε υπέρ της ε, Ανδρέα Μπότσκορ, της ε, υποψηφίου, με το κόκκινο κατά και με το άσπρο απέχουμε. Θα ήθελα να πω στα μέλη ότι σε περίπτωση που, γίνει, που ψηφίσετε λάθος μπορείτε να αλλάξετε την ψήφο σας μέχρι να κλείσω την ψηφοφορία. Τόσο χρόνο έχετε από τη στιγμή που ε, ξεκινάει η ψηφοφορία μέχρι τη στιγμή που κλείνει μπορείτε να αλλάξετε το κουμπί, να ξαναπατήσετε κουμπί για να αλλάξετε την ψήφο σας. Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε την ψηφοφορία. Ich frage, haben alle nach ihrem Willen abgestimmt? Ψήφισαν Πέρα τη ψηφοφορία. 15 υπέρ, 10 κατά, 5 αποχέ. Πρέπει να αφαιρέσουμε λοιπόν 5 ψήφου. Υπάρχει παρόλα αυτά η απαραίτητη πλειοψηφία. 25 ψήφοι. 30 ψηφίσαντες ψήφισαν ψήφου, έδωσαν ε, ψήφους 25, έχουμε 5 ε, που αφαιρούνται, οπότε 13 είναι η απαραίτητη ε, πλειοψηφία, οπότε γίνεται εξελέγει αντιπρόεδρος η κυρία Μποτσκορ. Θέλω να ευχαριστήσω τις πολιτικές ομάδες ε, που έτσι καταφέραμε να βρούμε μια λύση. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Αντρέ, ε, αγαπητή Ανδρέα, ελάτε εδώ στο βήμα. Έχουμε προβλέψει θέση για σας. Congratulations. So, ich darf nun mit feststellen, dass die Konstituierung Διαπιστώνουμε τώρα λοιπόν ότι η σύνθεση της ε, ομάδας ε, της Επιτροπής Πολιτισμού έχει κλείσει και πάμε στα διάφορα. Εδώ θα ήθελα σύντομα να πω, δεν έχουμε τίποτα για τη δημόσια συνεδρίαση. Οπότε να σας πω ότι στις 4 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα η επόμενη συνεδρίαση από τις 3 ε, μέχρι τις 6.30 και στις 5 Νοεμβρίου από τις 9 μέχρι τις 12.30 και από τις 3 μέχρι τις 6.30. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ παρά τις δύσκολες αυτές εποχές με τις ακροάσεις των Επιτρόπων και για την επικοδομητική σας συμβολή, συμβολή στην, Επιτρο... στην ακρόαση του Επιτρόπου Γκαμπριέλ χθες, της Επιτρόπου Γκαμπριέλ χθες το βράδυ. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας.